Εντάξει, σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. E, και σύμφωνα με το άρθρο 3, εδάφια 3 και 4, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στην συνεδρίασή της στις 11 ε, Απριλίου 2011 ε, επιβεβαίωσε τα διαπιστευτήρια του κυρίου Μπρουίς και προτείνει να κυρωθεί η εντολή του ήδη από τον Μάρτιο 2011. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, αντιρρήσεις, δεν βλέπω να υπάρχουν και έτσι η εντολή αυτή επικυρώνεται υπογραφή πράξεων νομοθετικού χαρακτήρα που αφορούν την κανονική διαδικασία που